τους στον κατάλογο ένα λεπτό ο καθένας. Ο λόγος στην κυρία Νίνα Τζίλ. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Ο κύριος Πόσπισιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να εξηγήσω την ψήφο μου για το ψήφισμα για το Ισλαμικό κράτος. Δεν ήταν ονομαστική η κλίση και θα ήθελα και οι ψηφοφόροι μου στην Τσεχική Δημοκρατία και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γνωρίζουν ότι ήμουν υπέρ του ψηφίσματος για το Ισλαμικό κράτος γιατί δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη μορφή μόρφωμα το Ισλαμικό κράτο, δεν θέλω να το αποκαλέσω κράτο, είναι μια ομάδα ανθρώπων που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και αυτό αποτελεί λοιπόν μια οργάνωση την οποία θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τώρα. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αξιολογούμε σωστά το κατά πόσο θα χρειαστεί να κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους. Γιατί αν δεν κάνουμε τίποτε, πολύ φοβάμαι ότι ο κίνδυνο του Ισλαμικού κράτους μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλε χώρε. Ευχαριστούμε. Δεν είναι εδώ ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να πω ότι καταψήφισα το ψήφισμα αυτό για το Ισλαμικό κράτος. Καταψήφισα μάλλον ε, και είμαι ενάντιο με το Ισλαμικό κράτο και υπερψήφισα βεβαίω το ψήφισμα. Δεν φαντάζομαι να είναι πολλοί βουλευτέ που δεν είναι υπέρ από το ψηφίσματο. Όμω αυτή την εξήγηση ψήφου θα ήθελα να επισημάνω ότι απαραίτητο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συμμαχοί τους θα πρέπει να δημιουργήσουν μια κοινή συμμαχία, μια μεγάλη συμμαχία με κοινή δράση κατά του Ισλαμικού κράτους βάσει της εντολής του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο που είχα την ευκαιρία να τονίσω, να δώσω έμφαση στην ανάγκη αυτή. Βεβαίως καταδικάζουμε το Ισλαμικό κράτος, ΕΣΑΗ, απλώς... Ε, τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμαχοί του ανά τον κόσμο θα πρέπει να βρουν την πυγμή για να αναλάβουν δράση κατά ε, τη περίπτωση αυτή. Δεν, δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουμε πολύ εύκολα από αυτό. Ε, ο κύριο Γιάρ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα το ψήφισμα και πρέπει να πω ότι συμφωνώ με όλα τα στοιχεία. Αλλά ήταν το σημείο 9 του ψηφίσματος με χαροποιεί όπου κοιτάζουμε και εν συντομία τις αιτίε. Η Ιρακινή κυβέρνηση καλείται να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτική στη σύνθεσή της και όλες οι πολιτικές ομάδες, όλες οι εθνοτικές ομάδες της κοινωνίας θα πρέπει να συμμετέχουν στην δίκηση και στην κυβέρνηση της Ιρακινής ε, διακυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτό ίσως να ήταν η γενεσιουργός αιτία που οδήγησε κάποιους ανθρώπους ε, στο ριζοσπαστικοποίηση και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι το ψήφισμα είναι ισόρροπο και θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε πλέον τα σημεία αυτά που αναφέρονται στην, ε, στο ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο λόγος τον κύριο Μπριουά. Δεν βρίσκεται στην αίθουσα, γι' αυτό θα ακούσουμε τον κύριο Κέλλη για να Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα είναι κρίμα που δεν είχαμε ονομαστική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία εδώ. Συνεπώς θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου καταδικάζουν επιφύλακτα τη δράση του Ισλαμικού κράτους μία από τις πιο βίες, τα πιο βία κινήματα που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Και οπωσδήποτε τη σύγχρονη εποχή όπου τόσες χώρες προσπάθησαν να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το να βλέπουν τις δραστηριότητες αυτού του Ισλαμικού κράτους με τους αποκεφαλισμούς, τη συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες, όλες ε, την αντιμετώπιση πολλών θεμάτων όπως τους αναγκαστικούς γάμους κτλ. που πρέπει ανεπιφύλακτα να καταδικάσουμε κάθε πράξη τους ε, και να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέθοδο για να βεβαιωθούμε ότι τέτοιες δραστηριότητες ε, δεν θα επαναληφθούν στην ιστορία μας στο μέλλον. σας ευχαριστούμε. Τα